Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Καθίστε παρακαλώ. Meine Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και άρχεται η συνεδρίαση. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόμορφη ε, δήλωση του καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας, τον κύριο Βέρνερ Φάιμαν, τον οποίο ορίζω. Καλώς ήρθατε κύριε καγκελάριο. Κυρίες και κύριοι, είδα κατά τη διάρκεια... Βλέπω εδώ πέρα πώς εκπροσωπείται η κυβέρνηση της Ισπανίας από τον ε, επί σειρά ετών στον κύριο Ινίγκο Μέντες Δεβίγκο, στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κύριε Καγκελάρια, σας ευχαριστώ για το ότι δεχτήκατε την ε, πρόσκλησή μου να έρθετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μιλήσετε με τους ε, βουλευτές μας για το πώς βλέπετε εσείς το μέλλον της Ευρώπης. Οπωσδήποτε το φέτος, το 2013, βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική φάση της ε, πολιτικής ε, στην Ευρώπη και χωρίς καμία αμφιβολία η συνοχή των λαών και των κρατών στην ε, κοινότητά μας, μια κοινότητα κρατών και εθνών, έχει αποφασιστική σημασία για το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το μέλλον, το οικονομικό, το οικολογικό και το νομισματικό και νομίζω πως πηγαίνουμε προς μια κατεύθυνση στην οποία εγώ και εσείς φαντάζομαι πριν από μερικά χρόνια δεν θα μπορούσατε να την είχατε φανταστεί. Η συζήτηση λοιπόν του κοινοβουλίου μας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με δηλαδή ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ταυτόχρονα επικεφαλής κυβέρνησης μιας κυρίαρχης χώρας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, πως σας ευχαριστώ που ήρθατε ως εδώ για να συζητήσουμε μαζί. Και θα ευχόμουν περισσότεροι συναδελφοί σας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ε, έρχονταν ως εδώ και να έκαναν διάλογο με τους ερετούς εκπροσώπους των λαών της ε, ευρωπαϊκής ε, κυβέρνησης από το να κάνουν ε, δηλώσεις ως εκπρόσωποι μιας χώρας στο έδαφος μιας άλλης χώρας. Και νομίζω πως θα συμφωνήσει μαζί μου και η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών. Τον λόγο τώρα έχει ο καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας, ο κύριος Φάιμαν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Χαίρομαι για το ότι βρήκατε το χρόνο να έρθετε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι μια ιδιαίτερη τιμή να παρευρίσκομαι εδώ και να συζητώ μαζί σας το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής μας κοινότητας. Σε μια στιγμή στην οποία πάνω από 5,5 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι είναι άνεργοι. Σε μια στιγμή κατά την οποία πάνω από 8,5 εκατομμύρια κάτω των 24 ετών δεν μπορούν να βρουν δουλειά, θα ήταν κοινικό να πούμε πως έχει περάσει η κρίση. Είμαι πεπισμένος όμως πως σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1930 έχουμε επιτύχει πάρα πολλά για να αντιδράσουμε συντονισμένα με προγράμματα επενδύσεων απέναντι σε αυτή την κρίση. Και η πρόβλεψη επίσης κάποιων πως ε, το τέλος, το τέλος του 2012 θα ήταν λιγότερες οι χώρες της Ευρωζώνης, όλοι αυτοί που προέβλεπαν την αποκάλυψη δεν επαληθεύτηκαν και αυτό χάρη στις κοινές μας προσπάθειες. Επιτύχαμε λοιπόν πάρα πολλά, όλοι μαζί, για τα οποία είμαι υπεπισμένος πως χωρίς την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ζημίες που προκάλεσε η οικονομική κρίση δεν θα είχαν αντιμετωπιστεί ε, όπως αντιμετωπίστηκαν. Βεβαίως δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι όσο είναι τόσο χαμηλή η ανάπτυξη και τόσο υψηλή η ανεργία. Εάν θέλουμε και εάν ενισχύουμε την Ευρώπη, ενισχύουμε τους εαυτούς μας. Εάν κάνουμε χειρότερη την Ευρώπη, ε, βλάπτουμε τους εαυτούς μας. Ε, θα ήθελα να το πω αυτό προερχόμενος από μια χώρα η οποία ανήκει στους λεγόμενους καθαρούς εισφορείς. Βεβαίω, όταν μιλάμε για καθαρούς εισφορείς, μιλάμε για το ότι αν μετρήσουμε τα όσα δίνουμε και τα όσα παίρνουμε από τον κοινοτικό προπολογισμό, φαίνεται πως δίνουμε περισσότερα. Αλλά δεν φαίνεται εκεί πέρα το πόσο εποφελούμαστε από τις εξαγωγές που κάνουμε και από το ότι πολλές αυστριακές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι πλέον έκτημα για μια χώρα και πρέπει να συνυπολογίζεται όταν κάνουμε απολογισμό των οικονομικών πλέον εκτιμάτων και μείων εκτιμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός βασικού κομματιού της, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μόνο λοιπόν μέσω αυτής της αλληλεγγύης που ούτως ή άλλως πρέπει να καθορίζει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα υπόδειγμα που σε αντίθεση με άλλες υπήρους ασχολείται με τη δημοκρατία, την ελευθερία αλλά και με τα κοινωνικά ζητήματα η αλληλεγγύη αυτή λοιπόν δεν μπορεί να περιορίζεται στα εθνικά σύνορα αλλά να επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη όλοι μαζί θα ευημερήσουμε ή θα δυστυχήσουμε. Και αυτό το λέω γιατί με ρωτάνε συχνά όπως και εσάς τι ε, έκαναν όλα αυτά τα μέτρα, οι ασπίδες προστασίας, ο μηχανισμός σταθερότητας, το δημοσιονομικό σύμφωνο, οι επενδύσεις που αποφασίσαμε, ο προϋπολογισμός, οι δημοσιονομικές προοπτικές ε, που ελπίζω πως θα συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια τι νόημα έχουν όλα αυτά, με ρωτάνε. Μπορούμε να απαντήσουμε με δύο τρόπους. Μπορεί κανείς να πει, κάτι για το οποίο είμαι επεπισμένος, όσον αφορά την κοινωνική συνοχή. Πως η κοινωνική ισορροπία οδηγεί σε αποδοχή από τον λαό και η ε, ιστορία έχει διδάξει πως οι γείτονες οι οποίοι στο παρελθόν πάλευαν με βία και πολέμους έχουν εντωμεταξύ δημιουργήσει μια κοινότητα στην οποία αποδίονται σε έναν ειρηνικό ανταγωνισμό και με ειρηνικό τρόπο επιλύουν τις διαφορές τους. Όταν λοιπόν ιδρύθηκε. Τότε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλβα οδηγηθήκαμε σε γενιές οι οποίες ε, ζουν πλέον σε ένα περιβάλλον ειρήνης. Βεβαίω έχουμε νέους οι οποίοι χάνουν την ελπίδα γιατί δεν βρίσκουν τι να κάνουν, γιατί τελειώνουν το σχολείο ή τις σχολές τους και δεν ε, μπορούν να ζήσουν από την δική τους εργασία. Γι' αυτό ακριβώς εδώ πέρα είναι κοινή μας αποστολή χωρίς εθνικά σύνορα η κοινωνική συνοχή. Αυτή δημιουργεί εμπιστοσύνη και μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε μια κοινή ειρηνική ανάπτυξη. Βεβαίως, σε πάρα πολλά απέχουμε ακόμα από αυτό φανταστούμε πως δεν είχαμε όλα αυτά τα μέσα στη διάθεσή μας. Ποιος θα είχε τότε βλαπτεί. Δεν θα ήταν αυτοί οι οποίοι κέρδισαν πάρα πολλά με την κερδοσκοπία, οι οποίοι απομακρύνθηκαν πολύ περισσότερο από την πραγματική οικονομία. Ποιοι είναι ε, αυτοί οι οποίοι πληρώνουν όταν χρεοκοπεί μια χώρα. Οι λάθος άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τα νοσοκομεία και τα φάρμακα και δεν υπάρχουν λεφτά γι' αυτά, πληρώνουν λοιπόν οι λάθος άνθρωποι γιατί οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ε, κερδοσκόπησαν πληρώνουν το λογαριασμό. Πρέπει λοιπόν από κοινού να φροντίσουμε να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα από την κρίση και σε αυτά ανήκει η οικονομία, η εξοικονόμηση, η ανταγωνιστικότητα, αλλά και οι ενισχυμένες επενδύσεις και η αλληλεγγύη. Γιατί βεβαίως περισσότερες επενδύσεις μπορούν να υπάρξουν ε, μόνο εάν οι χώρες έχουν την δυνατότητα γι' αυτό. Και ακόμα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά γι' αυτό. Καταπολέμηση της απάτης, της απάτης του ΦΠΑ, καταπολέμηση αυτών που προσπαθούν στη χώρα τους να μην πληρώσουν τους φόρους, δηλαδή καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Επίσης, ενίσχυση των φορολογικών αρχών, όχι μόνο να αποφασίζουμε δηλαδή φόρους στα χαρτιά, άρα να πληρώνονται κιόλας, κράτος δικαίου και άρα αξιοπιστία για τους επενδυτές Όλα αυτά μου φαίνονται πως είναι οι σωστές απαντήσεις. Οι σωστές απαντήσεις γιατί η πολιτική των περικοπών με τη μηχανή του γκαζόν, οριζόντια βλάπτει τη χώρα και στην αγοραστική δύναμη και στις επενδύσεις και στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση οι παράγοντες δηλαδή εκείνοι που κάνουν μια χώρα πιο ανταγωνιστική. Γνωρίζουμε πως έχει ασχεθεί πολύ κριτική αυτές τις μέρες και εβδομάδες και δημοσίως για τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Και αντιμετωπίζουμε πολλές τέτοιες ερωτήσεις. Αλλά είμαι πεπισμένος πως βεβαίω όταν είμαστε όλοι μαζί στην ίδια βάρκα δεν απολαμβάνουμε μόνο τον καλό καιρό, αλλά όταν η θύελα ταρακουνάει αυτή τη βάρκα, πρέπει όλοι να καταβάλουν προσπάθεια να πιάσουν το κουπί για να βγούμε ξανά σε ήρεμα νερά. Γιατί δεν επιτρέπεται να σταματήσουμε να διαχειριζόμαστε, όπως ε, λέω εγώ, τα χρέη. Γιατί όταν τα επιτόκια απέχουν τόσο πολύ όπως τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε η Γερμανία και η Αυστρία παραδείγματο χάρη έχουν τόκους ε, επιτόκια μακροπρόθεσμα κάτω από το 2% και αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση θα μας πληρώνουν και όλας όπως έγινε για α, ε, βραχυπρόθεσμα ε, ομόλογα που έφτασαν να μας πληρώνουν για να τα αγοράζουν. Και άλλες χώρες είναι στα επιτόκια 6, 7, 8% και έτσι υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση και κόστος σε αυτές τις χώρες και δεν υπάρχει η δυνατότητα για επενδύσεις. Είμαι πεπισμένος πως τα μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει είναι η αρχή μιας κοινή διαχείρισης των χρεών. Η διαχείριση των χρεών. δεν θέλω να παρεξηγηθώ εδώ πέρα όταν μιλάω για αυτήν. Δεν μιλάμε πως θα έχουμε ένα βαρέλι δίχως πάτο και θα έχει ευθύνη κάποιος άλλος για τα χρέη άλλου. Σημαίνει πως δεν θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο ή κερδοσκοπικές δυνάμεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ευρώπη. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της ιδέας ενός ταμείου εξόφλησης των κρατικών ομολόγων και μιας κοινή διαχείρισης των κρατικών ομολόγων, κάτι το οποίο θεωρούμε απολύτως σωστό. Εάν δεν μείνουμε μόνο στον τίτλο και μιλάμε για επενδύσεις, αλλά θέλουμε να δώσουμε πραγματικά τη δυνατότητα αυτής της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να σας ευχαριστήσω για το ότι και σε ζητήματα της επιτήρησης, της εποπτείας των χρηματαγορών μας στηρίξατε, όπως και στο ζήτημα του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα στην Αυστρία, το αποφάσισαν όλα τα κόμματα στο κοινοβουλίο μας και θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει τέτοιες ε, αποφάσεις ε, με μεγάλη πλειοψηφία. Αφενός πρόκειται για ένα σύμβολο πως και οι χρηματαγορές πρέπει να συνεισφέρουν όταν πρόκειται για την ε, απελευθέρωση κονδυλίων για να υπάρξει δυνατότητα ανάπτυξης στο μέλλον. Αλλά υπάρχει και ένας ρόλος φορολογικός. Έτσι ώστε οι υπηρεσίες και ειδικά οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ευρώπη να υπηρετούν την πραγματική οικονομία και όχι κάποια προϊόντα τα οποία κινούνται σε ένα καζίνο. Οπότε όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, η ρύθμιση, η επιτήρηση των τραπεζών, νόμοι περί χρεοκοπίας, όλα αυτά που πηγαίνουν προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας και βεβαίως υπάρχει και δίκαιη κατανομή του κινδύνου να μην επομίζεται ο ένας τον κίνδυνο και ο άλλος να πληρώνει το λογαριασμό. Όλα αυτά είναι ρυθμίσεις αναγκαίες για να δείξουμε στον λαό πως έχουμε ως, ε, μπορεί ως πολιτική υπεύθυνη να μην έχουμε όλα τα αναγκαία μέσα στη διάθεσή μας, αλλά μάθαμε πως χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα για να εγγυηθούμε στο μέλλον πως δεν θα επαναληφθεί τέτοια κρίση και πως πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Γι' αυτό τα μέτρα αυτά από το δίκαιο χρεοκοπίας των ε, τραπεζών μέχρι την ε, το διαχωρισμό πιστοτικών ε, και επενδυτικών δραστηριοτήτων και των λοιπών δραστηριοτήτων των τραπεζών είναι αναγκαία. Και άρα καταλήγουμε σε κάτι το οποίο εγώ θα έλεγα και αυτονόητο. Αλλά τελικά αποτελεί αντικείμενο μιας συζήτησης με διαφωνίες, αλλά θέλω να το τονίσω. Υπάρχει, εάν θέλετε, ένα ζήτημα κάποιας βασικής πρόνοια, κάποια βασικά ζητήματα στη ζωή, δηλαδή ενέργεια, άλλε υποδομέ ε, το πόσιμο νερό, όπου θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να προσπαθήσουμε να παραμείνουν σε κρατικά χέρια και να μην οδηγηθούμε σε λάθος δρόμους ε, απελευθέρωσης. Γιατί εύκολα πολλούνται αλλά δύσκολα ξαναέρχονται στα δημόσια χέρια. Και εδώ πέρα επίσης ισχύει αυτό το οποίο ζητάνε πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή οι πολιτικοί να ανακτήσουν τον πρώτο λόγο. Και η πολιτική με ήταν να ανακτήσει τον ε, πρώτο λόγο. Γιατί βεβαίως συχνά παρουσιάζονται οι πολιτικοί ως υπεύθυνοι. Γιατί δεν λένε την γνώμη τους για την κερδοσκοπία και για άλλα φαινόμενα. Και εδώ πέρα βεβαίως ανήκει και η απασχόληση των νέων μία εγγύηση κατάρτισης των νέων. Γιατί στην Αυστρία, ξέρετε, έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία και την χαμηλότερη ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία κατάρτιση ενός εξειδικευμένου εργάτη προσφέρει πάρα πολλά και στη βιομηχανία και η βιομηχανία στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι σημαίνει αυτό. Παίρνουμε ένα 16χρονο από τον δρόμο και του δίνουμε την δυνατότητα να εκπαιδευτεί σε ένα σύστημα το οποίο είναι διπλής εκπαίδευσης, εν μέρη στο σχολείο, εν μέρη στην επιχείρηση, πρακτικά, έτσι ώστε αργότερα να έχει μια δουλειά με υψηλή ε, ποιότητα, αλλά έχει και την ευκαιρία ο ίδιος να βγει ανεξάρτητος στην αγορά εργασίας το σύστημα αυτό διπλής κατάρτισης που έχουμε αλλά και η εκπαίδευση μιας θέσης, εγγύ, ε, μιας θέσης η εγγύηση μιας θέσης ε, κατάρτισης που δίνουμε είναι πάρα πολύ θετικό. Και θα πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους να μιλάμε για το τι θα κόψουμε και να πούμε πως θα επενδύσουμε όλοι όσοι ζητάνε επιστροφή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα επενδύσουμε στην κατάρτιση των νέων. πω θέλουμε να βγάλουμε ένα 16 χρονου 16χρονους, χρόνου να του πάρουμε από τον δρόμο και να βρεθούν σε μια θέση μαθητείας. Γνωρίζω πω ε, η Αυστρία έχει την ε, άποψη πως εάν πάρουν όλη η επιστροφή από τον κοινοτικό προπολογισμό πρέπει να την πάρει και η Αυστρία και βεβαίως ε, πέρα από τα αστικά κέντρα έχει σημασία και η ύπεθρος ε, και η αγροτική οικονομία για να φροντίσουμε πως αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει ως πολιτιστική και πολιτική ταυτότητα να διατηρηθεί. Και στα α, δύσκολα κομμάτια κοινά της γεωργίας, ε, π.χ στις απομακρυσμένες περιοχές ή όταν γίνεται βιολογική καλλιέργεια. Όλα αυτά πρέπει να ενισχυθούν στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε πολλά να συζητήσουμε ακόμα όσον αφορά τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, Αλλά ο στόχο πρέπει να είναι να κάνουμε κάτι θετικό στο τέλο να υπάρξει. Ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα για να ε, δείξουμε πως κάνουμε αυτό το οποίο απαιτούμε από τους άλλους, από τους επενδυτές στην οικονομία κτλ. Ότι δείχνουμε δηλαδή εμπιστοσύνη στο μέλλον της ευρωπαϊκής κοινότητας και στην αξιοπιστία της. Και να πω κάτι ακόμα για την αξιοπιστία αξιοπιστία και αηφορία στην ενεργειακή πολιτική είναι για μένα τον επικεφαλής αυστριακής κυβέρνησης ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρω βεβαίω πως για κάποιους αυτή η ενεργειακή αλλαγή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά η πυρηνική ε, ενέργεια δεν είναι αηφόρος πολιτική. Η πυρηνική ενέργεια τουλάχιστον από τη Φουκουσίμα και μετά έχει αποδειχθεί πως δεν μπορεί να ελεγχθεί. Θα δούμε και θα δούμε και στο μέλλον τι γίνεται και με την ενδιάμεση και με την οριστική διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων. Και αυτό νομίζω θα το δείξουν και τα stress tests ε, της ε, Κομισιόν αλλά εγώ είμαι πεπισμένος πως το ασφαλέστερο πυρηνικό εργοστάσιο είναι το εργοστάσιο που δεν υπάρχει. Ξέρω πως κάποιοι, βλέπω πως κάποιοι γελάνε. Οι άνθρωποι στη Φουκουσίμα όμω δεν έχουν καμία όρεξη για γέλια. Και είμαι πεπισμένο πως είμαστε εμείς η γενιά εκείνη η οποία θα απαντήσει σε κάποια χρόνια από σήμερα το ερώτημα το τι θα κάνουν οι επόμενε γενιέ με τα πυρηνικά απόβλητα. Και, ολοκληρώνω, είμαι υπερήφανο για τις γενιές που προηγήθηκαν, οι οποίες μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την εποχή της ανοικοδόμησης, βρήκαν το κουράγιο να οδηγηθούν σε αυτό το ειρηνικό έργο της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν υπολόγιζαν το τι γίνεται και αν αποδίδει και αν συμφέρει οικονομικά μήνα το μήνα αυτή η υπόθεση. Αλλά ήταν μια επένδυση στο μέλλον της χώρας. Και θα ήθελα να πω κάτι επίσης για την Νότια Ευρώπη. Αν κάποιοι σε κάποια χρόνια, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και από την Αυστρία, αλλά και παιδιά στην Ισπανία, στην Ελλάδα που μεγαλώνουν σήμερα, κρίνουν την σημερινή μας πολιτική, εγώ θα θέλω να μπορώ να τους πω το εξής. Η αλληλεγγύη και η αγάπη του πλησίων ήταν ισχυρότερη από την κερδοσκοπία και την απληστία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. ευχαριστούμε κύριε Καγκελάριο. Ο κύριος Μαρόζο για μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καγκελάριε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα σύντομα με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τον Καγκελάριο και τον πρόεδρο που οργάνωσαν αυτή τη συνάντηση γιατί η συνεργασία σε ενωσιακό επίπεδο είναι κάτι απαραίτητο αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Ο Καγκελάριος, Καγκελάριο Φάιμαν, με την επίσκεψή σας εδώ μας δείξατε ότι κατανοείτε ότι η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία πρέπει να ενισχυθεί και σε εθνικό και σε πανενωσιακό επίπεδο. Είναι γνωστή η δέσμευσή σας για την Ένωση και αυτά που είπατε σήμερα το αποδεικνύουν εκ νέου. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα την ευγνωμοσύνη μας αυτή να την επεκτείνω και στην κυβέρνηση και τη χώρα σας ολόκληρη. Διότι η Αυστρία υπήρξε ηγέτης στην εφαρμογή πρωτοποριακών ενωσιακών προγραμμάτων, ας πούμε τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που στην Αυστρία είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη. Η Αυστρία όπως ξέρουμε είναι η χώρα με, τον χαμηλότερο, με τη χαμηλότερη ανεργία των νέων. Επίσης σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας της ιδέας της εγγύησης νεολαίας. Επίσης υποστηρίζεται σε την ε, έγκριση σε ενωσιακό επίπεδο ενός ε, κειμένου για τα χρηματοπιστωτικά μιας συνθήκης. Και επίσης αναφέρω σε άλλο τομέα την δέσμευση της Αυστρίας για τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων και καθαρών πηγών ενεργείας ως το τη της καταπολέμησης των κλιματολογικών αλλαγών. Τέλος, θα ήθελα επίσης να αναφέρω την στήριξη της Αυστρίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Πυρηνική Ασφάλεια. Αυτά είναι απλώς παραδείγματα των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα σας για την Ευρώπη και ως πρόεδρος της Κομισιόν προσβλέπω σε συνέχιση της στενής μας συνεργασίας και ευχαριστώ την Αυστρία για τη δέσμευσή της στην Ένωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το λόγο Ζωζεφ Ντόλ. Αγαπητέ Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πέρασο, κύριε Καγκελάριε, κύριε Βέρνερ Φάιμαν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Καγκελάριο που παρουσιάστηκε εδώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υλοποιηθεί αυτή η συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα σας εκπλήξει ότι εμείς πιστεύουμε εδώ στην προστιθέμενη αξία της Ευρώπης που να έχει ένα αξιόπιστο προϋπολογισμό γιατί στα μέσα της οικονομικής κρίσης χάρη στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ορισμένα κράτη-μέλη μπόρεσαν να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους ε, και να μειώσουν το έλλειμμά τους η θεραλέα απόφαση που πήραμε αρχίζει να κραποφορεί στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ευρωζώνη κατορθώσαμε να μειώσουμε το χρέο ε, και νομίζω ότι πρέπει να το επενθυμίσουμε, να επενθυμίσουμε τι προσπάθειε που κατεβλήθησαν, αλλά επίση να μην ε, ξεχνάμε ότι πρέπει να ασκείται μόνιμη πίεση, δεν έχουν λυθεί όλα μας τα προβλήματα και όταν πιστεύουμε ότι η κρίση έχει μείνει πίσω μας, την έχουμε ξεπεράσει, αυτό θα προετοιμάσει τη δεύτερη κρίση και το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές σε πολλά θέματα αυτό. Και σήμερα, αν δεν ισχύει αυτό για την Αυστρία, ε, υπάρχει ψηλό επίπεδο ενεργείας στην Ευρώπη Ευρώπη, το υπενθυμίσατε, κυρίως ενεργεία των νέων. Σε πολλές χώρες ε, πάνω από το 50% των νέων είναι άνεργοι. Αυτό δεν είναι βιώσιμο και η απαραίτητη μεγέθυνση ε, για να δημιουργηθούν θέσει εργασία δεν έχει επέλθει ακόμα. Πρέπει να υπάρξει μια λύση για να βγούμε από την κατάσταση αυτή, να ενισχύσουμε την ένωσή μα. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη σε όλου του τομεί. Χρειάζεται περισσότερη εναρμόνιση. Και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το έλλειμμα τη Ευρώπη μα κοστίζει πολύ από κοινωνική σκοπιά με την απουσία κοινών κανόνων ε, για τις συντάξει, για την καταπολέμηση της ενεργείας, για την κοινωνική προστασία. Το να μην προχωρούμε σε αυτούς τους φακέλους είναι ότι θέτουμε σε κίνδυνο την ελληνική την ευρωπαϊκή από, από τη δημοσιονομική σκοπιά και μπορεί να δημιουργηθεί δημοσιονομικό dumping μεταξύ των κρατών. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να έχουμε τις ίδιες φορολογικές βάσεις ε, και για το ευρώ νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν είναι λογικό σε μια χώρα να μην υπάρχουν, ε, να υπάρχει κάποια ισχυρή φορολόγηση που και να κινητοποιεί τα άτομα και να προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού εναρμόνιση. Ε, δεν σημαίνει ταυτοποίηση, αλλά συνάδει με μεγαλύτερη διαφάνεια και από την τραπεζική σκοπιά ζητάμε ε, συχνά από την Αυστρία και το Λουξεμβούργο να θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία του 2003 για την αποτέμιευση ε, ορισμένοι ε, φοροδιαφεύγουν λόγω του τραπεζικού απορρίτου ε, και ξέρετε ότι η Αυστρία οφειλήθηκε πολύ από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αυστριακές επιχειρήσεις επενδύουν στις υποδομές στην Ευρώπη και αυστριακές τράπεζες είναι μεταξύ των πλέον δυναμικών ε, στην περιφέρεια. Όμως θα είχαν την ίδια επιτυχία αν δεν υπήρχαν κοινέ πολιτικές όπως ε, η πολιτική, η περιφερειακή πολιτική και η γεωργική πολιτική που παραδειγματικά έχει εφαρμόσει η Αυστρία και ε, εγώ όταν ε, μεταβαίνω ε, στην Αυστρία το βλέπω αυτό και κυρίως μην εγκαταλείψετε αυτές τις πολιτικές, ας δημιουργήσουμε και άλλες, αλλά μην εγκαταλείψετε αυτές τις πολιτικές γιατί θα υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Και επίση πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρώπη ε, είναι μία οδό διπλή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε αφενό να επωφελούμαστε από την ενία αγορά και από την άλλη σε περίοδο να αρνούμαστε να βοηθήσουμε όσου είναι σε δύσκολη θέση. Γιατί αυτό συνείσφερε στη δική σα επιτυχία και είμαι σίγουρο ότι θα αναλάβει η Αυστρία τι ευθύνε τη στο οικονομικό μοντέλο γιατί επωφελήθηκε από την έννοια αγορά. Γιατί όταν μια χώρα υποστηρίζει μια άλλη που προβαίνει στι απαραίτητε μεταρρυθμίσει, τελικά ενισχύει ολόκληρο το οικοδόμημα το να έχουμε αλληλοβοήθεια είναι σημαντικό, είναι θέμα αλληλεγγύης αλλά και ευθύνη και σήμερα δεν τίθεται θέμα αναδίπλωση στον εαυτό μας αντίθετα πρέπει να επενδύουμε, να κεφαλαιοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις και να χρησιμοποιούμε ως δυνατόν καλύτερα ένα πολιτή προϋπολογισμό. Αν ο καθένας ε, επενδύσει ένα σέντ ε, θα έχει και τα κατάλληλα ωφέλη αν υλοποιηθεί η ελληνική. Εμείς ξέρουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε σε εσά και σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Χάνες Πόμποντα. Ευχαριστώ, κύριε Καγκελάρια. Γνωρίζετε βεβαίως πως υπάρχει και το ρητό του ότι μαθαίνει κανείς πάνω στη δουλειά και εσείς πάνω στη δουλειά έχετε γίνει πολύ ε, φιλοευρωπαίος γιατί βεβαίως βλέπουμε πως μόνο μαζί μπορούμε να λύσουμε την κρίση και αυτό βεβαίως ε, ήταν προφανές για την Αυστρία γιατί βρίσκεται μεταξύ Ανατολής και Δύσης ε, Βορρά και Νότου αλλά βεβαίως όλοι ε, υποφέρουμε αν δείτε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία η φτώχεια και η ανεργία αυξάνονται. Δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι άρα για το ότι εμείς οι Αυστριακοί ή οι Γερμανοί είμαστε σε κάπως καλύτερη θέση. Πρέπει να έχουμε κοινωνικές δομές που δεν θα το ανέχονται αυτό. Και θέλω να υποστηρίξω αυτό το οποίο είπατε πράγματι για το ότι είναι απαράδεκτο αυτό το χάσμα, η ψαλίδα των επιτοκίων. Μιλήσατε για τα ευρωομόλογα και για το Ταμείο Εξόφλησης των Κρατικών Ομολόγων. Κάτι το οποίο εμεί συζητάμε ως Κοινοβούλιο και αναμένουμε από Συμβούλιο και Κομισιόν μια θετική απάντηση. Ή τουλάχιστον να σκεφτείτε πώς και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να συσταθεί ένα τέτοιο ταμείο. Γιατί ωραίο είναι να μιλάμε γενικά πως είναι πολύ υψηλή η ψαλίδα των επιτοκίων, αλλά πρέπει κάποια στιγμή και εσείς να το πείτε ξεκάθαρα και να το υποστηρίξετε. Και βεβαίως, κατά μία έννοια, η Αυστρία, θα μπορούσε κανείς να πει βεβαίως το λέει, πως το λέω επειδή είμαι Αυστριακός, και σοσιαλδημοκράτη. η Αυστρία είναι ένα ε, μοντέλο αντίθετο του νέου φιλελευθερισμού, πω η ανταγωνιστικότητα δηλαδή υπάρχει μόνο με την μείωση του κοινωνικού κράτους. Αντιθέτως εμείς αποδεικνύουμε πως το κοινωνικό κράτος και η ανταγωνιστικότητα πάνε χέρι-χέρι. Έτσι και είναι και πρέπει να είναι. Βεβαίω δεν είμαστε μια ε, ευτυχής απομονωμένη νήσος η Αυστρία, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική στάση της κοινωνικής εξίσωσης που οδήγησε προς τα εκεί. Και βλέπουμε πως ε, και η Γαλλία με τον πρόεδρο Ολάντα έδειξε πως είναι καλό οι κοινωνικοί εταίροι να αναζητούν ε, από κοινού λύσεις. Μιλήσατε για επενδύσεις. Οι ναι. επενδύσεις είναι δυνατές όταν δεν έχουμε μόνο μία πρωτόγονη πολιτική λιτότητας. Θα πρέπει να δούμε και την ε, πλευρά των εσόδων και όχι μόνο των δαπανών. Και βεβαίως την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Αυτό ζητάμε τώρα και για την Ευρώπη και όχι ως εθελοντικά μέτρα κάποιων χωρών. Όχι, πρέπει να είναι μια κοινή ευρωπαϊκή δράση και αυτό το οποίο προ την Κομισιόν είναι καλό, πρέπει να πάει ένα βήμα παραπέρα, πρέπει να διατηρηθούν και τα απαραίτητα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό αυτό ο προβολισμό. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για την εγγύηση για του νέου και να κόβουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όχι, θέλουμε περισσότερα λεφτά για να καταπολεμήσουμε την ε, των νέων. Φόρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ναι, γελάνε παντού και στη χώρα μου και στο εξωτερικό πάλι τα ίδια και πάλι με αυτό το φόρο. Τώρα ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποιο ε, θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ζητάμε τουλάχιστον από την Ιρλανδική Προεδρία. Αλλά κύριε Καγκελάρη θα με συγχωρέσετε γιατί βεβαίως το ανέφερε και ο κύριος Ντόλπος, και στο μέτωπο της φοροδιαφυγής χρειάζεται η συνεισφορά της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου να κάνουν κάτι θετικό σε αυτό το τομέα. Θα μπορούσε, παραδείγματο χάρη, η Αυστρία να διατηρήσει τραπεζικό απόρριτο για του Αυστριακού. Αλλά να υπάρξει υποχρέωση πληροφόρηση για του λοιπού. Για να υπάρξει ένα κοινό ευρωπαϊκό αγώνα κατά τη φοροδιαφυγή και να πιέσουμε και την Ελβετία για να δείξουμε πως και σε αυτή την περίπτωση και η Αυστρία και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση κινούνται από κοινού. Και τέλος, κύριε Καγκελάρια, αυτό το οποίο είπατε στα τελευταία σας λόγια. Εδώ και χρόνια πράγματι έχετε τραβήξει μια ξεκάθαρη γραμμή που σας διαχωρίζει από τον λαϊκισμό και την άκρα δεξιά. Τώρα για τον ε, λαϊκισμό δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Π.χ. αν ερχόταν εδώ πέρα και ο κύριος Κάμερον και έβγαζε τον ε, λόγο του που θέλει να βγάλει για την ε, Ευρώπη θα έβρισκε νομίζω αρκετούς εδώ πέρα να τον χειροκροτήσουν. Αλλά όσον αφορά τα ακροδεξιά κόμματα και ένα ξεκάθαρο όριο που πρέπει να υπάρξει είναι κάτι οπωσδήποτε που πρέπει να γίνει για την Ευρώπη και να το κάνετε δικό σας θέμα, δική σας υπόψη. Πρέπει να υπάρξει μία ενιαία γραμμή κατά τη άκρα δεξιά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και τώρα για τους φιλελεύθερους. Το λόγο έχει ο κύριος Φερχόφστοντ. Ευχαριστώ κύριε Καγκελάρη για την εμπνευσμένη ομιλία σας. Νομίζω καιρός ήταν να μιλήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης και είναι καλό που ακούσαμε κάποιον που προέρχεται από χώρα που είναι καθαρός εισφορέας που μας είπε τα επιχειρήματα που μπορεί να ισχύσουν έναντι κάποιου άλλου καθαρού εισφορέα από την άλλη πλευρά της μάχης. Βλέπετε ότι δεν έχουν την ίδια στάση όλοι οι καθαροί εισφορείς. Πρέπει να πω κύριε Φάιμαν, το είπατε κι εσείς, σε μια συνέντευξη πριν από μερικές μέρες, ότι μπορεί να υπάρξει κάποια σύγχυση ως προς το μέλλον της Ευρώπης από την άλλη μεριά της μάχης. Γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Κάμερον δεν συμφωνεί ούτε με τον εαυτό του για την ημερομηνία και τον τόπο της ιστορικής δήλωσης που θέλει να κάνει για το μέλλον της Ευρώπης. Βέβαια ιστορική θα είναι τον Παρασκευή η δήλωση για το μέλλον της Ευρώπης. Καλύτερα και από τη Θάτσερ στη Βρύγη. Την ξαναδιάβασα την ομιλία της στη Βρύγη. Ήταν πολύ φιλοευρωπαϊκή ομιλία. Είπε και το διαβάζω, διαβάζω τη Μάργαρετ Θάτσερ. πρέπει να κάνουμε περισσότερα όλοι μαζί. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζητάει ο κύριος Κάμερον και θα το ζητήσει, θα το δηλώσει την Παρασκευή. Πρέπει να πω όμως κύριε Πρόεδρε ότι σε αυτή τη συζήτηση και παρόντος του κυρίου Φάιμαν πρέπει να απαντήσουμε στον κύριο Κάμερον ότι ήδη ξέρουμε τι θα πει την Παρασκευή. Νομίζω ότι εξ ονόματος της πλειοψηφίας εδώ μέσα μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει θέμα για μεμονωμένη ατομική από μία χώρα μέλος ε, αναδιαπραγμάτευση. Ούτε από τη Βρετανία ούτε από άλλη χώρα. Για έναν απλό λόγο. Χρειαζόμαστε μία ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κάρτο όπως συμβαίνει σήμερα με εξαιρέσεις, με απαλλαγές, με επιστροφές αυτό που σκοτώνει την Ένωση σήμερα είναι αυτή ακριβώς η προσέγγιση. Υπάρχει η αρχική Ένωση των 6, υπάρχει η Ένωση των 12 που είναι το ελάχιστο που χρειάζεται για να εφαρμοστεί το χρηματοπιστωτικό συμβόλαιο. Υπάρχει η Ένωση των 17, η Ευρωζώνη, η Ένωση των 25 με το Σέγγεν και η ολόκληρη Ένωση των 27. Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι είναι πολύ περίεργο είδο ζώου η Ένωση. Μερικές χώρες μέλη δεν υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα, ενώ άλλες και εκτός από την Ένωση καλούνται να συμμετάσχουν. Η Ελβετία είναι τμήμα του Σέγγεν. Η Βρετανία όμως τμήμα της Ένωσης δεν ανήκει στο Σέγγεν. Πώς το εξηγούμε αυτό στους πολίτες, αυτή την Ευρώπη à carte, όπου καθένας διαλέγει ό,τι θέλει. Αναδιαπραγμάτευση λοιπόν από το Ηνωμένο Βασίλειο ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν θα μπορούσε παρά να χειροτερέψει τα πράγματα. Επίσης πιστεύω ότι μια τέτοια ένωση αλακάρτ όπως γίνεται τώρα, όπως θα μας πει ο κύριος Κάμερον την Παρασκευή, μόνο να σκοτώσει μπορεί την ενιαία αγορά, ο καθένας μπορεί να επιλέξει τι θα μείνει από την ενιαία αγορά, αν παραδείγματο χάρη οι Γάλλοι πουν μα «Ε, μας αρέσει μεν η βιομηχανική πολιτική αλλά όχι οι κανόνες του ανταγωνισμού ή αν πούν οι Γερμανοί μας αρέσει η ενιαία γερμανοι μα αγαθών αλλά όχι υπηρεσιών. Τι θα μείνει από την ενιαία αγορά. Ας είμαστε ειλικρινεί και να είναι ειλικρινεί και ο κύριο Κάμερον. Μία αναδιαπραγμάτευση όπω θέλει σημαίνει μάλλον το τέλος της ενιαίας αγοράς ίσως και της ένωσης ολόκληρης. Και αυτό συνάδελφοι δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών ούτε των Βρετανών διότι δεν μπορεί να οδηγήσει παρά σε αυτή την κατάργηση της ενιαίας αγοράς ή σε κάποια δευτερεύουσα σχέση με την Ένωση και τη Βρετανία όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, χώρες που πληρώνουν αλλά δεν έχουν λόγο και θα ήταν ανόητο για μια χώρα με 53% των εξαγωγών της στην Ένωση. Και ακόμη πιο είναι τόσο ανόητο ώστε και οι καλύτεροι φίλοι της Βρετανίας, οι Αμερικανοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Καταλήγω λοιπόν κύριε Πρόεδρε δεν θέλουμε ατομική μεμονωμένη αναδιαπραγμάτευση για να μειώσουμε ό,τι κοινό έχουμε. Θέλουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτά που ζητάει ο κύριος Κάμερον και θα μας τα πει την Παρασκευή. Χρειαζόμαστε μια κοινή προσπάθεια για να καθοριστεί μια πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη γιατί αν θέλουμε κύριε Φάιμαν να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα και τις προκλήσεις που δίκαια αναφέρατε στην ομιλία σας τότε μόνο με μια πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και όχι με μονομένα με αναδιαπραγματεύσεις από μία ή άλλη χώρα μέλος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους. Τον λόγο έχει η κυρία Ρεμπέκα Χάμς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, κύριε Καγκελάριε. Πρέπει να παραδεχτώ πως τις τελευταίες ημέρες ε, προετοιμαζόμενοι για αυτή τη συζήτηση χάρηκα για τις ε, εξελίξεις ε, και τις θέσεις σας για την Ευρώπη. Κοιτάξαμε με θαυμασμό την Αυστρία και χαιρόμαστε για το ότι βλέπουμε τέτοια δυναμική παρουσία υπέρ μιας κοινή ευρωπαϊκής λύσης της χειρότερης κρίσης που ζούμε εδώ και χρόνια. Και εγώ διάβασα αυτή την συνέντευξη που ανέφερε ο κύριος Φερχόφστατ και θεωρώ το ότι θεωρώ πως όλοι πρέπει εδώ πέρα να συνυπογράψουμε τη δήλωσή σας πως το πρόβλημα του χρέους που αφήσαμε να αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λυθεί από κοινού και να επανέλθει η πρόταση του Ταμείου Εξόφλησης των Χρεών, βεβαίως όχι υπό όρους ε, ρόδινους, αλλά είναι μια πρόταση που σωστά έκαναν οι λεγόμενοι σοφοί της οικονομίας και είναι νομίζω ένας δρόμος βατός Επίσης, στο άρθρο σας βρήκα δηλώσεις ε, που λένε πως πρέπει να είναι υπομονετικός κανείς στην Ευρώπη και πως τα πράγματα διαρκούν περισσότερο από όσο θα θέλαμε. Θεωρώ πως μία λύση αρχής του ζητήματος του χρέους δεν πρέπει να καθυστερήσει πάρα πολύ γιατί αλλιώς τα πράγματα οξύνονται και στον κοινωνικό τομέα κατά το οποίο περιγράψετε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Είπατε στη συνέντευξή σας πριν έρθετε εδώ πέρα πως η Ευρώπη δεν πρέπει να επιτρέψει την ε, όξυνση της κοινωνικής ανισότητας και αδικίας. Αυτό όμως γίνεται ήδη. Αν θέλετε η Ευρώπη συνολικά να έχει περισσότερα κονδύλια για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, αυτό πρέπει να το τονίσετε και εδώ μέσα και ε, εκτός, κατά το οποίο κάνετε βεβαίως, αλλά τότε πρέπει να συνταχθείτε με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό και τις ε, μεσοπρόθεσμες ε, δημοσιονομικές πρόπτικες. Η ομάδα μου θεωρεί ανησυχητικό το ότι πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση της μη μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής χωρίς το πρασίνισμά της προς μια αλλαγή. Επίσης βρίσκουμε απειλητικό το ότι τα ταμεία συνοχής δεν θα αλλάξουν και ταυτόχρονα χωρίς αλλαγή της γεωργικής πολιτικής, χωρίς αλλαγή των διαρθρωτικών ταμείων ε, επιχειρείται περικοπή του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει πως όλα τα φιλόδοξα καινοτόμα σχέδια, είτε είναι η εγγύηση για τους νέους, είτε οι άλλες καινοτομίε για την κοινωνική ισότητα, δεν θα είναι πλέον δυνατά. Έχουμε έναν προϋπολογισμό της Ευρώπης προ-νεωτερικό, χτεσινό. Θα πρέπει να τα πείτε αυτά τα πράγματα, να μπει δυναμικά η Αυστρία στην συζήτηση του προϋπολογισμού. Η Αυστρία αποτελεί ε, υπόδειγμα. Δόξα το Φίσλερ, μπορώ να το πω σήμερα αλλά το πρασίνισμα που πρότεινε ο Επίτροπος ε, Τσόλος δεν ε, μπορεί να γίνει και χωρίς να ε, αλλάξει κάπως η κατάσταση και δεν έχουν να φοβούνται τίποτα οι αγρότες της Αυστρίας και αλλού. Τώρα για την πυρηνική ενέργεια, πολύ καλά όλα αυτά τα οποία είπατε για την πράσινη ομάδα, τα τεστ κοπόσεως ε, οριστικοποιήθηκαν παρά τις προσπάθειες ε, του κυρίου Έτιγκερ και βεβαίως υπάρχει και η οδηγία για τις προδιαγραφές ασφαλείας για την ευθύνη σε πυρηνικά ατυχήματα, πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής είναι κενές υποσχέσεις. Και εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να κινηθείτε πιο δυναμικά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύρια Χάρμς για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς, ο κύριος Κέλνεν. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καγκελάρια, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κύριου Φερχόφστατ. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο να σταθούμε σε αυτό το θέμα Μίλησε ε, τόση ώρα για μια ομιλία που δεν έχει καν ακούσει του Ντέιβιτ Κάμερον. Αλλά εντάξει, βελτιώνονται τα πράγματα. Δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να τσιτάρει την Μάργαρετ Θάτσερ με θετικό τρόπο. Θα σας στείλω ένα βιβλίο με ρίσεις της Μάργαρετ Θάτσερ στο μέλλον, εάν θέλετε. Είναι σημαντικό όμω να έχουμε μια, σημαντική, μια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη, μια συζήτηση όπου θα διαφανεί το πραγματικό επίπεδο, η κλίμακα τη κρίση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται μονάχα για να θεραπεύσουμε την κρίση του ευρώ. Απλώ να καταλάβουμε ότι στον παγκόσμιο στίβο, τον οικονομικό στίβο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα τα οποία απειλούν το μέλλον μα. Θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα την, το γεγονό ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανησυχία στην κοινή γνώμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο για την κατεύθυνση που ακολουθούμε δεν φτάνει να πούμε ότι ο κόσμος έχει άγνοια ή να πούμε ότι όλα αυτά είναι λαϊκισμός. Αν οι πολίτες έχουν σταματήσει να εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι πολλοί από του ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σταματήσει να εμπιστεύονται του πολίτε τη Ευρώπη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Χρειαζόμαστε μια νέα κατεύθυνση για την Ευρώπη. Πιστεύω, πιστεύω ότι θα πρέπει να αρθρώσουμε ένα νέο μήνυμα το οποίο να αποτελεί μια νέα κατεύθυνση για την Ευρώπη. <clears throat> Θέλουμε να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή συνεργασία, αλλά αυτό σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε εκβάθρον τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Γιατί βρίσκεται στο, στο σταυροδρόμι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ελέγχθη, το μοντέλο αυτό της ε, όλο και πιο στενής ένωσης απέχει τόσο πολύ από αυτά τα οποία θέλουν οι πολίτες και μπορούν να αντέξουν οι οικονομίες μας που Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο μοντέλο, όχι μια εσωστρεφού ολόπιε πιο έντονη ένωση, αλλά μια ένωση η οποία είναι πρακτική και εύκαμπτη. Πώ μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, Μπορούμε καταρχήν να ανοίξουμε τι αγορέ μα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την γραφειοκρατία και το βάρος της. <clears throat> Μπορούμε να προχωρήσουμε πίσω άμα καταλάβουμε ότι το κράτος έθνος δεν είναι κάτι το ξεπερασμένο, αλλά είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της σωστής διακυβέρνησης. Μπορούμε να πάρουμε λοιπόν μια λογική αντιμετώπιση για όλα τα προβλήματά μας και όχι να επιτρέψουμε η ιδεολογία να καθορίζει την πορεία μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημεία κίνηση. Μπορούμε να σκεφτούμε και πάλι όλο το ενωσιακό εκτιμένο και τις ρυθμίσεις οι οποίες επιβαρύνουν τις αγορές μας και χάνουν θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε μια πολιτική δράση για να δώσουμε νέα στεναρότητα στην ενιαία αγορά με την ψηφιακή οικονομία. Να μπορέσουμε να επανεξετάσουμε όλο το προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να έχουμε πραγματικά προσθέμενη αξία στην ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη και να αλλάξουμε ρυθμό στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τι ΗΠΑ, την Ινδία και άλλε αναδυόμενε οικονομίε που είναι αυτέ οι οποίε έχουν το δυναμικό ανάπτυξη και μπορούν να το δώσουν και στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά μπορούν να γίνουν δυνατό αν σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι εμεί έχουμε ω πολιτική τη λύση σε όλα τα προβλήματα. Πέραν τη Μάργαρετ Θάτσερ, εγώ μπορώ να σα παραθέσω τον Ρόναλτ Ρέγκαν και είπε ότι οι πιο τρομακτικέ ε, ένωση της αγγλικής γλώσσας είναι ότι θα πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι εδώ να σας βοηθήσω. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τους ανθρώπους να αναλάβουν την ευθύνη για τις δράσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Αν θέλουμε να έχουμε μια ισχυρά οικονομική Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβουμε το καλύτερο που μπορούν να κάνουν οι πολιτικοί είναι να σταματήσουν να αποτελούν εμπόδιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καγκελάρη, η Ευρωκρίση έχει δημιουργήσει μια έχει σπάσει τη συνένεση ότι μπορούμε να συνεχίσουμε όπως έχουν τα πράγματα. Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο, όχι μια Ευρώπη à la ούτε μια Ευρώπη με πρώτη και δεύτερη κατηγορία μελών, αλλά ένα εύκαμπτο, ευέλικτο μοντέλο το οποίο να συγκλίνει γύρω από την εσωτερική αγορά, όπου η κάθε χώρα μπορεί να συμβάλλει επί τη βάση των συμφερόντων τη και των αναγκών τη. Μια ένωση όπου όλα τα κράτη-μέλη είναι πράγματι σεβαστά και όπου υπάρχει πραγματική ένωση στην πολυμορφία. Ευχαριστώ κύριε Κάλανεν για την ε, Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, ο κύριος Χέλμερ. Κύριε Πρόεδρε, ο Καγκελάριος φαίνεται ότι κατανοεί κάποια από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η λύση γι' αυτόν είναι η περισσότερη Ευρώπη. Αυτό αποτελεί τον θρίαμβο της ελπίδας ε, έναντι της πείρας, ε, της προκατάληψης έναντι της καθημερινότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι σε μακροπρόθεσμη πτώση, ύφεση. Το 1998 ήταν περίπου 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ ο προπολογισμό τη Ένωση. Σήμερα είμαστε στο 20%, μέχρι το 2050 μπορεί να είμαστε στο 10% ή ακόμα και λιγότερο, ενώ αποφασίσουμε να παραμείνουμε στου στόχου για τη μείωση των εκπομπών, που σημαίνει ότι θα κατακαιρματίσουν την αγροτική οικονομία. Κύριε Φερχώστατ, σα πειράζει να μιλήσω. Ο λόγος λοιπόν για αυτή την πτώση δεν είναι ε, καλά καθορισμένος. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τελωνιακή ένωση, αλλά οι τελωνιακές ενώσεις είναι ένας παροχημένος ε, ε τρόπος εργασίας του 19ου αιώνα και μάλιστα κανείς ε, άλλος στον κόσμο δεν χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, η Τελωνιακή Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει ε, υπερβολική ρύθμιση και πάρα πολλούς κανονισμούς. Οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις ε, στοιχίζουν 100 δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο και αυτό μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τρίτον, υπάρχει μια ενεργειακή πολιτική η οποία δίνει στην Ευρώπη την πιο δαπανηρή ενέργεια παγκοσμίω. Αυτό υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητά μα και ε, υπάρχουν ε, ε, επιχειρήσεις παράκτιες οι οποίες παίρνουν τους ανθρώπους μα ε, στο εξωτερικό και οδηγούν τον κόσμο στην ε, ένδια χωρίς να καταφέρουν να μειώνουν τις εκπομπέ υποθηκεύετε τις ε, ζωές των παιδιών μας και των εγγονών μας κυρία Καγκελάρια και ε, τέλος έχουμε την καταστροφή του ενιαίου νομίσματος όπου ένας ε, Βρετανός καγκελάριος το αποκάλεσε την πιο ανεύθυνη περιπέτεια του, της μεταπολεμικής εποχής ο κύριο Μπαρόσο λέει ότι το χειρότερο της κρίσης πέρασε. Μην το πιστεύετε. Τίποτα δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες μεταξύ Δύσης, ε, ε, Βορρά και Νότου. Θα χρειαστούν και άλλες διασώσεις, θα χρειαστούν μόσιμε, ε, μόνιμες, μακροπρόθεσμες ε, εισρωέ χρημάτων από το βορρά στο νότο και αυτό δεν θα το δεχτούν οι Γερμανοί φορολογούμενοι και θα οδηγήσουν στη λιωτότητα και στην ανεργία που προσπαθείτε να λύσετε στην ε, ε, Νότια Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και να διασπαστεί. Υπάρχει ήδη μια πολιτική για την Δημοσιονομική και Τραπεζική Ένωση που δημιουργεί διαιρέσει και δημιουργεί πρόβλημα μεταξύ της Ευρωζώνης και των υπολόπων. Στη χώρα μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει ολοένα αυξανόμενη αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Πρωθυπουργό νομίζει ότι θα μπορέσει να τη μειώσει αυτή την αντίθεση ζητώντα εκ νέου χώρε των αρμοδιοτήτων. Ε, αλλά οι πολίτε έχουν καταλάβει ότι το αν ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι είμαστε λιγότερο δημοκρατικοί και λιγότερο ελεύθεροι. Όλοι ζητούν ανεξαρτησία, δημοκρατία, ελευθερία και όσοι το αναζητούν πολύ καλά κατάλαβαν ότι καλύτερα θα ήταν να μείνουμε απ' έξω. Ευχαριστώ. Για την Ενωμένη Αριστερά έχει το λόγο η κυρία Τσίμα. <coughs> Κύριε Φερχόφστατ, αφήστε με. Κύριε Φερχόφσταρτ, ίσως θέλετε να ακούσετε και αυτά που θα πει η κυρία σήμερα. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται προκλήσεις όπως έχουν γίνει από την απέναντι πτέρυγα. Κύριε Καγκελάρια, θέλω να σας εκφράσω την... το σεβασμό μου και τη χαρά μου για την έλευσή σας. Έχετε τονίσει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι δεδομένο ότι τα μέλη του, Συμβουλίου θα, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έρχονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να λάβουν μέρος στις συζητήσεις. Το έπραξε αυτό η κυρία Μέρκελ τον προηγούμενο Νοέμβριο, αλλά ένα χελιδόνι δεν φαίνει την άνοιξη. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν και μεγαλύτερη κατανόηση από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν φλιαρεί απλώς για τα θέματα αυτά. Μόνο από κοινού μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί το Συμβούλιο να βρει τις σωστές λύσεις με απόλυτο σεβασμό για τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ακούγοντας και τα α, επιχειρήματα του Κοινοβουλίου ακόμα και αν είναι αντίθετα από αυτά τα οποία έχει το Συμβούλιο. Παραδείγματο χάρη το θέμα του πολιετούς, των πολιετών δημοσιονομικών ε, προοπτικών το να μειωθούν αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εγώ κατανοώ όλα αυτά τα οποία είπατε εδώ σήμερα σαν μια προσφορά αλλά και σαν μια έκκληση προς τα άλλα μέλη του Συμβουλίου να κινηθούν και να ακολουθήσουν την κατεύθυνση αυτή. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια στάση απόστασης εναντί της ιστορινής κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωση που γίνεται διακριτική αντί να ακολουθεί την ενωσιακή μέθοδο και επίση, δεν πιστεύουμε ότι η λύση είναι να αναχθεί η δημοκρατία στις οικονομικές σχέσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και να κατανοήσουμε ότι έχουμε μια ευθύνη για έναντι των ανθρώπων σε οποιαδήποτε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μονάχα τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλους αυτούς που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι πολίτε είτε είναι μετανάστες ή πρόσφυγες ή οτιδήποτε τέτοιο, όλοι αυτοί έχουν δικαιώματα τα οποία πρέπει να γίνουν σοβαστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοηθήστε μας να συμβάλλουμε στο ότι μελλοντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα εξακολουθήσουν να είναι σοβαστά σεβαστά και να μην περιοριστούν μονάχα στο δικαίωμα να ασκεί κανείς ελεύθερα εμπόριο και δραστηριότητες οικονομικές στην εσωτερική αγορά. Εφέτος είναι το έτος των Ευρωπαίων πολιτών δεν πρέπει να χάσει το περιεχόμενό του. Μας ενδιαφέρει να είναι σαφές τους ε, πολίτες ότι έχουν δικαιώματα όχι μονάχα μέσα στην εσωτερική αγορά αλλά και ευρύτερα. Πρέπει να ξαναστήσουμε στα πόδια της τη δημοκρατία και οι πολίτες της Ευρώπης να μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτή και να ξέρουν ότι γίνεται ακουστή η φωνή τους. Η δημοκρατία και η δημοκρατικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επίτευξη της αλληλεγγύης, η οικοδόμηση μιας κοινωνικής ένωσης στην Ευρώπη, όλα αυτά είναι αλληλένδετα θέματα. Σας ζητώ λοιπόν και σας ζητώ και από όλους τους άλλους στο Συμβούλιο, α σταματήσει αυτή η πολιτική λιτότητος ακόμα στην Ευρωπαϊκή στη ζώνη του ευρώ. Ακόμα και η Κομισιόν έχει παραδεχθεί ότι αυτή η πολιτική λιτότητα δεν είναι ο τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον οποίο θα μπορέσουμε να βγάλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από την κρίση. Από την κρίση. Καταλάβετε ότι δεν μπορούν να συνεχίζουν τα πράγματα έτσι ώστε να ξεπουλούνται οι δημόσιοι πόροι και να ιδιωτικοποιούνται. Όλα αυτά είναι εναντίον της ύπαρξης ενός μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μεγαλύτερη αλληλεγγύης. Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης και αποκρατικοποίησης καταλεί τις δημόσιες παροχές και αρχές. Η ιδιωτικοποίηση του συστήματος κοινωνικών παροχών, η έλλειψη ελάχιστου κοινωνικού επίπεδου προστασίας και ελάχιστο επίπεδου περιβαλλοντικής προστασίας στρέφεται εναντίον όλων των Ευρωπαίων. Εάν πραγματοποιηθούν αυτές οι απειλές, τότε δεν θα υπάρξει μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πούν δεν θέλουμε μια τέτοια ένωση πια. Δεν θέλουμε λοιπόν να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα τέτοιο σημείο που να την απορρίψουν οι ίδιοι οι πολίτες της. Θα πρέπει για να μην συμβεί κάτι τέτοιο να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον θα πρέπει οι δημοσιονομικές προοπτικές να βρίσκονται σε ένα επαρκές επίπεδο. Είναι παράλογο να υπάρχουν κόμματα στην Bundestag τα οποία είναι έτοιμα να καταψηφίσουν για προγράμματα τα οποία είναι προγράμματα βοήθειας. Αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά. Σας ζητώ λοιπόν να υπάρξει μια πραγματική υποστήριξη για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που σοβεί στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Τσίμερ. Για τους μη εγγεγραμμένους έχει το λόγο ο κύριος Χάνς Πέτερ Μάρτιν. η πρακτική της κριτικής μας έχει φέρει σε ένα σημείο το οποίο δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ακόμα περαιτέρω αντιπαραθέσεις. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία ανέφερε ο Καγκελάριος στον λόγο του. Πράγματι υπάρχουν στοιχεία που θα πρέπει να επικρίνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως το οποίο χρειαζόμαστε στην κρίση αυτή είναι να βρούμε κάποιες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο πολυδιάσπασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Καγκελάρη, μιλήσατε για την αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Το παρελθόν όμως, η αλληλεγγύη αυτή ήταν περισσότερο με τις τράπεζες, υπερβολικά μαζί με τις τράπεζες και ελάχιστα με τους πολίτες. Δεν πρόκειται για την αντιμετώπιση μόνο των χρεών βλέπουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το χρέος το κρατικό, είναι η δύναμη των τραπεζών. Είναι το λεγόμενο too big to fail, ότι οι τράπεζες έχουν υπερβολική δύναμη και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Έχουμε τη σκιώδη τραπεζική διαδικασία η οποία διακινεί κολοσιαία ποσά. Βλέπουμε ότι τα χρέη καταλήγουν στις κεντρικές τράπεζες και δεν, και δεν βοηθούν να εξασφαλίσουν τις τράπεζες. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να σκεφτείτε την πραγματική συμμετοχή των πολιτών, ώστε να έχουμε μια ένωση των πολιτών και όχι μονάχα μια τραπεζική ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Καγκελάρη, παρακαλώ. Θα κατανοήσετε ίσως ότι εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση μέχρι στιγμής, χωρίς να πω τώρα σε λεπτομέρειες σε αυτά που έλεγχαν. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε δύο σημεία, τα οποία μέσα σε αυτό το ε, σύντομο διάστημα που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να τα αναφέρω. Καταρχήν για αυτά που είπε ο κύριος Κάλανεν για την ευελιξία. Η ευελιξία για κάτι το οποίο δεν είναι δίκαιο είναι αρνητική. Η, η ευκαμψία με τη δικαιοσύνη μαζί είναι κάτι το θετικό. Και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα με ποιο τρόπο θα μπορέσει να ενταχθεί αυτή η ευελιξία στο οικονομικό μας σύστημα. Έχει νόημα να κάνουμε τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση των δομών και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει εξοικονόμηση με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει η ευελιξία αν ορισμένοι αναλαμβάνουν κινδύνους και σπεκουλάρουν οι τραπεζίτες και ο χρηματοπιστωτικός κύκλος και τελικά την ύφη να την πληρώνουν οι απλοί φορολογούμενοι. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα πλαίσιο κανόνων που να εξασφαλίσουν την ισοδίκαια μεταχείριση. Όταν καθένα παίρνει κάποιε αποφάσει, θα πρέπει να επομίζεται αυτό τον κίνδυνο των αποφάσεων αυτών. Επομένω, είτε κάποια εποπτικά συμβούλια στι τράπεζε ή κάποια νομοθεσία για την αφαιρεγκαιότητα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτή η αλληλεγγύη, ότι αυτή συγγνώμη, η ευελιξία λειτουργεί με τρόπο ισοδικαίο για όλου. Και θα ήθελα να σταθώ στον κύριο Χέλμερ. Ο κύριο Χέλμερ αναφέρθηκε στην αντίθεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα του. Αυτό έχει νόημα μονάχα όταν θέλει αυτό το κράτος να σπρώξει όλα τα στραβά στο καλάθι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει για τον εαυτό του να κρατήσει όλα τα επιτέγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονάχα. Λοιπόν, εκεί πρέπει να υπάρξει πραγματικά και μια βελτίωση και σε επίπεδο εθνικής πολιτικής και όχι μονάχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν πρέπει να συνεχίσει αυτή η απόθεση των σφαλμάτων και του φτεξίματος στους άλλους. Σε αυτά που είπε ο κύριος Φροχοστάτ προηγουμένως, έχουμε αυτή τη στιγμή αυτά που είπε ο κύριος Κάμερον, τα οποία έχουν δημιουργήσει πολλές αντιπαραθέσεις. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε εμείς να ενισχύσουμε τις χώρες μας ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερο σε επίπεδο αγοράς. Εάν όλοι κάνουν το δικό τους τμήμα θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε. Και τέλος το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας το οποίο αναφερθήκαν. Μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα εάν δώσουμε στους νέους μια καλύτερη κατάρτιση και μια καλύτερη δυνατότητα να εργαστούν. Γι' αυτό υποστηρίζω την εγγύηση για τους νέους. Μπορούμε να αυξήσουμε λοιπόν επίσης την ανταγωνιστικότητα αν είμαστε καινοτόμοι. Αυτό είναι δύσκολο, το ξέρουμε όλοι. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε αρκετούς πόρους για έρευνα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις δύσκολες εποχές είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν πόροι για αυτή την κατεύθυνση. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να ενισχυθεί με το να έχουμε μια κοινή προσπάθεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχουμε και την ανταγωνιστικότητα που έχουν άλλες χώρες του κόσμου με μεθόδους που ε, δυστυχώς δεν είναι πάντα δημοκρατικές. Δεν πρέπει να απανηθούμε όμως το δικό μας μοντέλο της δημοκρατίας και της ελευθερίας στο βωμό της ανταγωνιστικότητας. Το μοντέλο αυτό δεν λέει ότι θα πετύχουμε την ανταγωνιστικότητα με το να μειώνουμε τους μισθούς και τις κοινωνικέ παροχές. Αυτό είναι ασύμβατο με το δημοκρατικό μοντέλο της Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό θα χάσουμε την υποστήριξη των λαών μας και γι' αυτό είμαι απόλυτα υπερήφανο, γιατί εμείς μπορούμε να αγωνιζόμαστε για την ανταγωνιστικότητα διατηρώντας το δημοκρατικό μοντέλο της Ευρώπης. Ευχαριστούμε κύριε Φάιμαν. Ερχόμαστε τώρα στου ομιλητέ από τι πολιτικέ ομάδε Ο κύριος Καράς έχει το λόγο. Κύριε Καγκελάρια, κύριε και κύριοι, είναι σημαντικό το ότι σήμερα είστε παρόν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμείς χαιρετήσουμε ιδιαίτερα αυτό το μήνυμα που δίδετε ως αρχηγός κράτους προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας λέω λοιπόν ότι χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς ως ε, καγκελάριος μπορείτε να μιλάτε <clears throat> για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας το κάνουμε και άλλοι είτε υπέρ είτε κατά. Η Αυστρία λόγω της γεωγραφικής της θέσης και λόγω της ιστορίας της είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με την ανάπτυξη και την συνέχιση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Γι' αυτό σας ζητώ Κάντε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε το ταχύτερο δυνατό να μπορέσει να υπάρξει η συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική ένωση. Δεσμευτείτε στο μέλλον να σταματήσουν οι κεκλεισμένων των θυρών διασκέψεις κορυφών, κορυφής. Και ας περάσει το Συμβούλιο στο επίπεδο ενός δεύτερου νομοθετικού σώματος όπως και το Κοινοβούλιο. Ενώπιον της κρίσης και της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αποφασιστικό τρόπο στο επόμενο βήμα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πιο ανοιχτή και ουσιαστική διαβούλευση με τους πολίτες. Η Αυστρία, λόγω της ιστορικής της εμπειρίας, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, έχει στηρίξει ιδιαίτερα το κοινωνικό μοντέλο. Ήταν και ένας από τους μοχλούς ολοκλήρωση στην Ευρώπη και θα πρέπει να είναι και ένας μοχλός στην μελλοντική ολοκλήρωση και διεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο στόχος θα πρέπει να είναι η Ευρώπη να είναι και στο μυαλό αλλά και στην καρδιά των πολιτών. Δεν θα πρέπει λοιπόν η αντιμετώπιση του προπολογισμού να αντιμετωπίζεται με τη λογική πληρώνω λιγότερα και θέλω να πάρω περισσότερο. Έχει αναφερθεί το θέμα των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη γεωργία. Δεν φτάνουν όμως όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει όλα τα κονδύλια που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να φέρει σε πέρα στους στόχους και τα εγχειρήματα που ζητούν από αυτήν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ένα ακόμα σημείο για το θέμα του δημοψηφίσματος. Πρέπει η ευρωπαϊκή διάσταση και η ευρωπαϊκή ευθύνη που έχει επέναντι στο διεθνή κόσμο να είναι και αυτή ορατή στα θέματα αυτά. Η ευρωπαϊκή λοιπόν συνειδητοποίηση θα πρέπει να αναδημιουργηθεί. Θα πρέπει να έχουμε μια νέα συνένεση ώστε οι πολίτες της Ευρώπης να μπορούν να θεωρούν ότι είναι τμήμα μιας κοινότητος και δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι τα παιχνίδια τα οποία παίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι μονάχα παιχνίδια εθνικών εγωισμών που στρέφονται εναντίον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ήτανε λίγο, ήμουνα λίγο γενναιόδωρος, διότι επρόκειτο για ένα αυστριακό ομιλητή. Για τους άλλους ίσως μπορώ να περικόψω λιγάκι το χρόνο. Θα είμαι γενναιόδωρος μόνο με τους αυστριακούς. Έχουμε καθυστέρηση λιγάκι. Ο κύριο Λάιφρυντ τώρα, ο οποίο είναι γνωστό για την ικανότητά του να παραμένει στα χρονικά όρια. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Πάντα προσπαθώ. Ο κύριος Χέλμερ μίλησε για καταδαπάνηση κοντιλίων. Αλλά νομίζω ότι ένας καλοπληρωμένος ευρωβουλευτής θα πρέπει να σκέφτεται λίγο περισσότερο προτού μιλάει για τέτοια θέματα χθε, πριν έρθει ο κύριο Καγκελάριο, μου είπε ένα Ιταλό συνάδελφο, καλό είναι που έρχεται ο κύριο Φάιμαν. Γιατί είναι απαραίτητο στο Συμβούλιο κάποιο να μιλήσει για τα κοινωνικά θέματα και να τονίσει τη σημασία του. Σημασία των. Δεν είναι τόσο απλό βέβαια, είναι δύσκολο το να ξέρουμε τι θα πρέπει να κάνουμε, γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό το ότι ήρθατε εδώ να εκφράσετε αυτή την άποψη. Όταν πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε προσπάθειες για την αλληλεγγύη, για την ισότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μονάχα όχι σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Αλλιώς θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η ανεργία των νέων στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα χειρότερο από το να έχετε νέου οι οποίοι δεν έχουν καμιά προοπτική, κανένα μέλο. Νέοι οι οποίοι είναι πολύ καλά καταρτισμένοι και μορφωμένοι, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα και είναι στον δρόμο, δεν έχουν απολύτω τίποτα. Αυτή την πρόκληση λοιπόν δεν μπορούμε να την αφήσουμε να είναι έτσι. Στην Αυστρία έχουμε βρει τρόπου να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Αυτέ οι λύσει μπορούν να λειτουργήσουν και από κοινού στην Ευρώπη. Μπορούμε στην Ευρώπη όλοι μαζί να βρούμε τρόπου να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων και να δώσουμε στου νέου μια προοπτική για το μέλλον. Με αυτή λοιπόν την κοινή θέση δεν αρκεί να συζητάμε. Θα πρέπει να μπορέσουμε να πετύχουμε και την συμμετοχή των πολιτών της Ευρώπης, να δώσουμε ενθουσιασμό στους νέους της Ευρώπης. Για να μπορέσει λοιπόν να διατηρηθεί αυτή, αυτός ο ενθουσιασμός για την Ευρώπη θα πρέπει να στραφούμε έναντι αυτών που είναι κατά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Που λένε πετάξτε την τάδε χώρα έξω γιατί δεν έχει πάει καλά στα οικονομικά της. Γιατί δεν πληρώνουν οι πολίτες τους φόρους τους ή οτιδήποτε τέτοιο. Η καταστροφή του ευρώ θα ήταν μεγαλύτερη καταστροφή στην Ευρώπη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Δεν είναι το πρόβλημα που θα θίξει μονάχα δεν θα θίξει του κερδοσκόπου, θα θίξει του απλού ανθρώπου οι οποίοι υποστηρίζουν την Ευρώπη. Και πιστεύω κύριε Καγκελάριο, με αυτά τα οποία είπατε βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτό το οποίο μπορούμε να πετύχουμε από κοινού είναι πολύ περισσότερο από το αριθμητικό άθροισμα των επιτυχιών που μπορούν να έχουν τα κράτη-μέλη μας αριθμητικά και μεμονωμένα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας κατευθύνει στις μελλοντικέ ενέργειες που θα κάνουμε για τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάιφρυντ. Για τους φιλελεύθερους το έχει το λόγο η κυρία Βέρτμαν. Κύριε Καγκελάρια, η παρουσία σας σήμερα με κάνει να ελπίζω ότι θα υπάρξουν και άλλοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που θα έρθουν εδώ για να συζητήσουν μαζί μας και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα είναι πάρα πολύ καλή για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αυστρία έχει μια ιδιαίτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω σε αυτά που είπατε για την αντιμετώπιση της ανεργία και της ανεργία των νέων. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ακόμα ένα πολύ ψηλό επίπεδο ένδυας στην Ευρώπη. για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ανεργία και η ενεργεία των νέων, θα πρέπει να γίνουν τα κατάλληλα βήματα, τα οποία όμω θα έχουν ένα αηφόρο χαρακτήρα. Και έρχομαι εδώ πέρα στην ε, δική σας ε, πρόταση να μειωθούν οι επιστροφές, να, να διαγραφούν μάλλον οι επιστροφές του προϋπολογισμού σε όλους. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποδεχθούμε ότι οι νέοι μας εξακολουθούν να είναι άνεργοι παρά την καλή τους κατάρτιση. Όταν βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο πλοίο, θα πρέπει όλοι από μαζί να κατευθύνουμε το πλοίο προς την ίδια κατεύθυνση, όχι ο καθένας από εκεί που θέλει. η κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε, πρέπει να είναι η σωστή, η βιώσιμη κατεύθυνση και μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κεκτημένα 60 ετών ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούνατσεκ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Καγκελάρια. Και εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και τη χαρά μου που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσετε μαζί μου, χωρί καμία ηρωνική διάθεση. Σα έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα οποία έχετε τονίσει και στο παρελθόν ω Ευρωπαίος και ω τμήμα του κυβερνητικού συνασπισμού τη ε, Αυστρία. Νομίζω λοιπόν ότι και η σημερινή σα ομιλία είναι προ την ίδια κατεύθυνση. Είναι απαραίτητο να υπάρξει σεβασμός για την κοινωνική Ευρώπη. Η εγγύηση αυτή για τους νέους που συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα με πρωτοβουλία των πλασίνων είναι ένα σημαντικό σημείο. Όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι όμως, αυτή η εγγύηση για τους νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτεί περισσότερα χρήματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτά τα χρήματα, γιατί όταν μιλάμε για χρήματα θα πρέπει να επανέλθω σε εσά και να ζητήσω από την Αυστρία να συμφωνήσει σε μια, σε μια γενική συμφωνία κατά της φοροδιαφυγής και να μπορέσει να διακόψει συμφωνίες όπως παραδείγματος χάρη με το Λουξεμβούργο που επιτρέπουν σε ξένους φοροφυγάδες να θέτουν τα κονδύλια τους σε τράπεζες όπου δεν κινδυνεύουν να φορολογηθούν. Αυτό ζητώ από σας λέει κύριε καγκελάριο. Επίση, ένα δεύτερο στοιχείο. Βρισκόμαστε σήμερα στο Στρασβούργο. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρει έδρε. Πριν από τρει μήνε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει με μεγάλη πλειοψηφία να ζητήσει από το Συμβούλιο να ακολουθήσει ένα κοινό σχέδιο μαζί μα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ μια ενιαία έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε εξοικονομίε. Θα ήθελα και πάλι να σα παρακαλέσω να προωθήσετε αυτή την πρωτοβουλία στο Συμβούλιο, να δείτε ποιο είναι το κόστο αυτή τη ύπαρξη τριών εδρών και να μπορέσουμε να καταλήξουμε καιρό σε μια μοναδική έδρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την ομάδα της Ελευθερίας της Δημοκρατίας, ο κ. Πάξας. Καγκελάριο Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα είναι κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για την ενωμένη Ευρώπη όπου ισότιμα κράτη συνεργάζονται. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε διότι ο Δάλος οι προσδοκίες μας να γίνουμε μια ισχυρή και ανεξάρτητη κοινότητα τελικά θα μας διαιρέσει διότι κάποιοι θα θελήσουν να υπερισχύσουν και θα θέλουν να είναι κάποια κράτη εξαρτημένα από την βούληση και τις αποφάσεις των ισχυροτέρων κρατών. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινότητα ίσων κρατών ε, αλλά να μην ισχύει πραγματική ισότητα. Ε, κλειδονίζεται η Ένωση από την ανεργία και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για βασικά πράγματα όπως την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζω ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη η κοινότητα των κρατών και όσο περισσότερο μιλάμε για την ομοσπονδικοποίηση και την απελευθέρωση τόσο όλο ένα και περισσότερο θα θέλουν να φύγουν. Ο κύριος Μέλτσερ από Υπάρχει όλο και μεγαλύτερο σκεπτικισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και η έννοια ανασφάλεια, ακόμα και απόρριψη. Πάρα πολλοί είναι αγανακτισμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταμαρτυρούν το δημοκρατικό έλλειμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ και είναι πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα τη Ευρώπη, αλλά μάλλον ομφαλοσκοπεί. Εμεί θέλουμε να υπάρξει καλύτερη προσπάθεια πληροφόρηση, η οποία να καταδεικνύει και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά στοιχεία <clears throat> τη παρουσίες των χωρών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά δεν προέρχονται από μένα, δεν προέρχονται από κακούς δεξιούς λαϊκιστές. Αυτά είναι στοιχεία που έχουν ε, δημοσιευθεί και έχουν συζητηθεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και σε άλλες χώρες. Όταν λοιπόν έχει κανείς μια αντιμετώπιση η οποία αφήνει όλα αυτά τα προβλήματα να πλανώνται, θα πρέπει να δεχθεί την ε, καταγγελία και τις επικρίσεις. Θέλουμε, θέλετε κύριε Καγγελέα να ακολουθήσετε το συμφέρον του αυστριακού λαού ή των γραφειοκρατών. Ο κύριος Κέλαμ για το ΕΛΚ έχει τώρα το λόγο. The future of Europe. Πρόεδρε, το μέλλον της Ευρώπης σημαίνει κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τις βασικές πολιτικές μας διότι η επιλογή δεν είναι ανάμεσα στην Ομοσπονδιακή Ευρώπη για την Ευρώπη των Εθνών, είναι ανάμεσα στην υπεροχή των κοινών συμφερόντων ή των εθνικών και βραχυπρόθεσμων συμφερόντων. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλιση, η κοινή αμυντική πολιτική, η κοινή ενεργειακή πολιτική, η κοινή πολιτική για την κυβερνοασφάλεια και η ολοκλήρωση πάνω απ' όλα της ενιαίας αγοράς ε, και η ολοκλήρωση της οικονομική και νομισματικής αυτό είναι το πραγματικό μέλλον τη Ευρώπη και δεν είναι ε, σε καμία περίπτωση ουτοπία. Μπορούμε να το πετύχουμε. Είναι πρόβλημα πολιτική βούλησης. Αυτή έχει εκλείψει, αλλά όχι μόνο. Είναι ένα πρόβλημα νοοτροπίας επίσης. Κοιτάζουν τα κράτη προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και θεωρούν ότι είναι εταιρείε που πρέπει να τους παρέχουν υπηρεσίες. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος. Μπορεί να θεωρήσουμε ότι είμαστε συνειδιοκτήτες και του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως συνεπάγεται και κοινή ευθύνη και όχι μεταφορά και μετακύληση ευθυνών προς τους ερετούς εκπροσώπους των λαών ή τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά να κάνουμε όλη μια προσπάθεια να αλλάξουμε ίδιοι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έδειξαν ε, τουλάχιστον ε, δύο πράγματα. Πρώτον, η οικονομική κρίση βασίζεται σε μια βαθιά ηθική κρίση, κρίση αξιών. Δεύτερον, ε, ότι το μοντέλο ευημερία και κράτου πρόνοια των τελευταίων δεκαετιών δεν θα είναι πλέον βιώσιμο και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η αλλαγή τη νοοτροπία, χρειάζεται να επομεστούμε όλοι τι ευθύνε μα. Είναι κέρια σημασία γιατί νομίζω ότι όσα θα καταρρεύσουμε όλοι μαζί. Η κυρία Μπέρε, τώρα από πλευρά των ε, σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καγκελάρια, για τα κοινωνικά ζητήματα η Αυστρία αποτέλεσε τη βάση μια πολύ καλή πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την πρωτοβουλία για την νεολαία. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό λοιπόν ε, που μπορέσ... Ε, σας ευχαριστώ που μπορέσαμε να ακολουθήσουμε αυτό το στόχο μέχρι τώρα και ελπίζω ε, στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ στο Δουβλίνο η πρόταση αυτή να γίνει πλέον ευρωπαϊκή πρόταση ώστε στους τέσσερις μήνες που θα ακολουθήσουν, που θα είναι μια δύσκολη κατάσταση για τους νέους, να καταφέρουμε να βρούμε μια λύση και η λύση που έχετε προτείνει ε, να πόκειται βασικά στη ε, κινητοποίηση των κοινωνικών κονδύλων της Ευρώπης και ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να προτείνετε ε, να έχουμε ένα 20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όλα αυτά στα πλαίσια του προπολογισμού, το οποίο θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε αυτή την αλληλεγγύη, την οποία ε, μας είπατε ότι επιθυμούμε να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να επιτύχουμε αυτή την αλληλεγγύη θα πρέπει οι Έλληνες, για παράδειγμα, να μπορέσουν να νοικοδομήσουν την φορολογική τους βάση. Και εδώ ο ε, κύριος που ήρθε να μαζί δει τις προάλλες μας είπε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα ε, είναι δύσκολη διότι οι Γερμανοί θεωρούν ότι ε, ε, πληρώνουν οι ίδιοι την κατάσταση για την Ελλάδα. Θέλουμε λοιπόν την οδηγία για την ε, φορολογία και θεωρώ ότι η στάση σας είναι κρίσιμη για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη αλληλεγγύη και να έχουμε τη δυνατότητα ένα κράτος όπως η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την αλληλεγγύη και να μπορέσει να υπάρξει αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τους μία έχει τώρα το λόγο ο Κύριε Καγκελάρια. η αντιμετώπιση της κρίσης ήταν πολύ σημαντική στη χώρα σας. Το ερώτημα όμως είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει με την κρίση. Έχουμε ουσιαστικά μετακυλήσει τον κίνδυνο στους Ευρωπαίους ε, φορολογούμενους. Δεν έχουμε λύσει κανένα πρόβλημα. Έχουμε εξαγοράσει μόνο με μερικά δισεκατομμύρια την διάσωση. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα ανεργίας των νέων που πλησιάζουν ή ξεπερνούν το 50%. Έχουμε καταλήξει σε μηδενική ανάπτυξη. Έχουμε θέσει σε κάποιο βαθμό από κοινού τα χρέη μας. Έχουμε τροφοδοτήσει την κερδοσκοπία δεν υπήρξε κάποια συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις ζημίες οι οποίες προεκλήθησαν παρά το γεγονός ότι το είχαμε ε, υποσχεθεί στους Ευρωπαίους φορολογούμενους, δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου σε επίπεδο φορολογικής δικαιοσύνης, όταν να το κάνει αυτό ο κύριος Ολάντ, τον κατήγγυλαν και τον καθίβρισαν όλοι. Έχουμε λοιπόν χώρες οι οποίες παίρνουν χρήματα χωρίς να έχει προκύψει καμία απόλυτα διαρθρωτική τροποποίηση και χωρίς να έχει υπάρξει εξυγίανση των ε, οικονομικών τους. Απλώς είπαμε ότι τώρα πάνε όλα καλά. Με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Για την ομάδα του ΕΛΚ, ο κύριος Μίλαν Μον έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Καγκελάρη για το πνεύμα αλληλεγγύης και για τις ε, σκέψεις που μας παρουσιάσετε για το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο ε, σήμερα δεν είναι τόσο αβέβαιο όσο πριν από ένα χρόνο το Συμβούλιο ε, και τα όσα αποφάσισε στο δεύτερο εξάμεινο του 2012, καθώς ε, και οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μας επέτρεψαν να διασκεδάσουμε λίγο τις αμφιβολίες και για το ευρώ και για τη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Αλλά τα όσα επιτύχαμε δεν αρκούν. Θα πρέπει να γίνουν και εθνικέ μεταρρυθμίσει, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να προοδεύουμε ώστε η οικονομική και φορολογική ένωση να, και δημοσιονομική συγγνώμη, ένωση να συνεχιστεί και ε, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από την κρίση. Ε, στο λεγόμενο έγγραφο των τεσσάρων προέδρων θα πρέπει να το στηρίξουμε και είναι γνωστή η στήριξη των Ισπανικών αρχών προς αυτό. Κύριε Καγκελάρη, εγώ θεωρώ ότι η κοινή γνώμη και όπως είπατε και εσείς οι νέοι στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική. Αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να βοηθήσει την κρίση και αν θεωρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λύση και όχι πλέον το πρόβλημα. Αυτό είναι αυτό το οποίο νομιμοποιεί σήμερα την ε, Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτά είναι τα μέτρα για να διαφύγουμε τις κρίσεις. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο ενός ε, πολύπλευρου κόσμου ε, όπου τα πάντα είναι αλληλεξαρτώματα. Και όπω μα υπενθύμισε ο Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Μπαρόζο, το μέγεθο μετράει και εμεί ενωμένοι θα είμαστε ισχυροί. Αλλιώ θα είμαστε άσχετοι. Και το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο ενοποιημένη εξωτερική πολιτική όπω μας ζήτησε άλλωστε και η συνθήκη τη Λισαβόνα. Για του σοσιαλιστέ, ο κ. Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καγκελάρια, η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης σημαίνει ότι απαντούμε σε δύο ερωτήσεις. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι πόρος ή είναι καταβόθρα της ανάπτυξης και η ανάκαμψή του μπορεί να επαφίεται μόνο στα κράτη-μέλη ή θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πραγματική δημοκρατική κυβέρνηση του ευρώ. Η απάντησή μας ε, είναι θετική από πλευρά τη ομάδα μας και στις δύο και χαιρόμαστε που τα όσα ακούσαμε από εσά οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μια Ευρώπη της σταθερότητας, της ανάπτυξης, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Το να ξεπεράσουμε την ε, ε, τυφλή λιτότητα δεν σημαίνει ότι θα ξαναγίνουμε ανεύθυνοι ε, από δημοσιονομική άποψη. Θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκέ πολιτικέ οι οποίε θα καθορίζονται σε συναπόφαση για την ε, κοινωνική ανάπτυξη και γι' αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό αντάξιο του ονόματό του που θα βασίζεται σε ένα ταμείο μείωση του χρέους και εκτίμησα ιδιαίτερα τα όσα άκουσα από εσά και μία ε, δημοσιονομική εξηγήση που θα είναι φίλος τη ανάπτυξη και θα βοηθά τις κατάλληλε πολιτική και δεν θα τιμωρεί τι δημόσιε επενδύσει. Γι' αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε έναν ισχυρό κοινωνικό πυλώνα, ο οποίος θα ξεκινά από την ενίσχυση τη ευρωπαϊκής εγγύησης για τους νέους, ε, όπου στην Αυστρία λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά. Κύριε Καγκελάρη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και τα όσα μας είπατε. Είμαι βέβαιος ότι από εδώ και πέρα, στους επόμενους μήνες, ε, η μάχη για την καθορισμό μιας κοινωνικής συμφωνίας και μιας πραγματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης θα βασίζεται και στη στήριξή σας. Κύριο το λόγο για το ΕΛΚ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την ευρωπαϊκή σας δέσμευση, καγκελάρια, αλλά περίμενα περισσότερα για την μελλοντική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική από το καγκελάριο μιας χώρας ε, ε, που είναι ως ε, σάντουιτς ανάμεσα στη, στα νέα και στα παλιά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε πολύ κοντά στα νέα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ε, πώς επιτοπλίστων δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη και δεν είπατε τίποτα για τον κίνδυνο της Ευρώπης δύο ταχυτήτων και για την απειλή που υπάρχει να διχοτομηθεί και πάλι η Ευρώπη. Νομίζω ότι για την Αυστρία που παραδοσιακά υποστήριζε τις ε, χώρες της ε, Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και την Κεντροανατολική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πει περισσότερα πράγματα. Ε, δεν θα έπρεπε να χαλάσουμε την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων γιατί αυτό είναι εις βάρος των συμφερόντων της Αυστρίας. Μιλούσατε, μιλήσατε στην αρχή της παρέμβασής σας ε, για τις ε, χώρες που καθαρά συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό. Δεν μου αρέσει να το λέμε αυτό, διότι εννοούμε ε, τις πλούσιες χώρες. Συγγνώμη, αλλά οι πλούσιες χώρες έχουν επωφεληθεί από ολόκληρο τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Δεν θα πρέπει μέσα στο συνταγματικό μας σύστημα να ενσωματώσουμε διαιρέσεις τέτοιου τύπου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να αλλάξει το ειδικό βάρος προς το κέντρο Ευρώπη ε, και ε, με φυγόκεντρε δυνάμει, σε βάση των οποίων ε, κάποια κράτη θα απομακρυνθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουμε απορρίψει προτάσει για την συστασία επίσημη επιτροπή όπου θα συσκέπτονται μόνο τα μέλη τη Ευρωζώνη και θα φασίσουν για τον προπολογισμό. Σα ευχαριστούμε και ο κύριο Μπρόκ από πλευρά του ΕΛΚ εν τέλει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καγκελάρια, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μακρύς ο δρόμος ο οποίος έχει, μας έχει φέρει ως εδώ με όλους αυτούς τους λόγους, αλλά ήταν ένας σωστός δρόμος, ένας θετικός δρόμος και ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία τόνισε ο κ. Καγκελάριος για την ε, εξυγίανση των οικονομικών, την μεταρρύθμιση των δομών στα πλαίσια πάντα μιας κοινωνικής Ευρώπης. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να ακούσουν αυτά τα λόγια όλοι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να συνεδριάσουν τον επόμενο μήνα για, την, ε, για τις ε, πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές να μην στραφούν εναντίον των στόχων της καινοτομίας και της πρόοδου της Ευρώπης. Η εσωτερική αγορά και η πραγματοποίηση της πλήρους εσωτερικής αγοράς σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να δεχθούν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια βάρη. Αυτό δεν είναι αυτό το οποίο είπε ο Ντέβιτ Κάμερο στην ομιλία του της ε, Παρασκευής. Επίσης το ευρώ δεν μπορεί να είναι το νόμισμα των 25, πρέπει να είναι το νόμισμα των 27. Δεν μπορεί να υπάρξει opt-out στα θέματα του ευρώ και της Οικονομικής Ένωσης, ούτε της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Δεν πρέπει με τον τρόπο αυτό να καταστραφεί η ενότητα της Ευρώπης, γιατί όλα αυτά θα έχουν αρνητική επίπτωση στο μέλλον. Και θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτά τα οποία είχε πει ο Ζαν Μονέ για την ενότητα της Ευρώπης. Ο καγκελάριος Φάιμαν έχει το λόγο κύριε Πρόεδρε. Για μια φορά ακόμα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την διενέργεια αυτής της συζήτησης. Επιτρέψτε μου μια μικρή επίκριση που δεν στρέφεται στο μεγαλύτερο μέρος των, των Ευρωπαίων ε, κοινοβουλευτικών. Είναι φανερό ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, όπως φάνηκε και στη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι ήταν παρόντες σε αυτή τη συζήτηση, γιατί θεωρώ μια συζήτηση με τον κύριο Σέσελ δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα όσο μια συζήτηση με τους ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους αυτούς που πήρανε τον κόπο να έρθουν εδώ σε αυτήν την ε, συζήτηση και είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμή για μένα να με προσκαλέσετε κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία ιδιαίτερα. Πρώτα απ' όλα, ο διχασμός της Ευρώπης. Και εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ιδίω μια χώρα όπως η Αυστρία, η οποία είναι πολύ καλά, στενά συνδεδεμένη με τις νέες χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτιστικά και ιστορικά και οικονομικά έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη όπως αναφέρθηκε για να εξασφαλίσει την ενότητα της Ευρώπης. Γι' αυτό δεν θέλουμε να υπάρξει διχασμός της Ευρώπης, να καταλήξουμε σε μια Ευρώπη η οποία θα έχει δύο ταχύτητες ή δύο κατηγορίες κρατών και είναι απαραίτητο για κάτι τέτοιο να διατηρήσουμε μια ενιαία Ευρώπη με ένα ενιαίο νόμισμα. Αυτή όμως η Ενωμένη Ευρώπη δεν θα πρέπει να έχει τη μορφή που διαγράφει για αυτήν ο Ντέβιτ Κάμερον. Για να έχουμε μια ενιαία ε, Ευρώπη με μία ταχύτητα δεν σημαίνει ότι ο ένας θα πρέπει να μένει ακίνητος και να εμποδίσει τους άλλους να προχωρήσουν. Αν θέλουμε λοιπόν όλοι να κινούνται με την ίδια ταχύτητα, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο χώρος των οικονομικών και των χρηματοπιστωτικών θα πρέπει να τύχει περαιτέρω συζήτηση, αλλά δεν θα πρέπει να παραμείνει το μόνο μας εγχείρημα. Θα πρέπει να είναι ένα τμήμα μονάχα της συνολική πρόοδου. Θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να υποστηρίξουμε τις ε, επενδύσεις, να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, να δώσουμε εγγύησει στους νέους. Γι' αυτό πρέπει προηγουμένω να επιτύχουμε αποτελέσματα στον οικονομικό χώρο, στα δημοσιονομικά μα και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κινηθεί για τα θέματα αυτά θα πρέπει και αυτοί να κάνουν κάποιες προσπάθειες να βγουν από την ακινησία τους γιατί αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό για τους πολίτες της Ευρώπης. Θα πρέπει να υπάρξουν πια αποφάσεις για την Ευρώπη οι οποίες θα καταδείξουν ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τους είναι σε θέση να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά. Έχουμε ευθύνη να δώσουμε μια απάντηση στις αιτήσει των πολιτών. Και θέλω να σταθώ τώρα σε αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Στάτλερ. Για ένα λεπτό, σκεφτείτε κύριε Στάτλερ. Ας, είχαμε, ας πούμε ότι είχαμε αφήσει κάποιες χώρες να χρεοκοπήσουν τα προηγούμενα χρόνια. Τι θα είχε προκύψει. Ίσως κάποιοι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων οι οποίοι είχαν κερδίσει πολλά στην κρίση πριν από την κρίση, αυτοί θα είχαν πληγεί από την χρεοκοπία αυτή. Όχι, θα είχαν πληγεί οι απλοί πολίτες οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθεια και την υποστήριξή μας και αυτό θα είχε καταστρέψει την ελπίδα για τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Θα είχαν πάψει να πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει ένα κοινό μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό εγώ είμαι υπερήφανος για το ότι καμία χώρα δεν αφέθηκε να χρεοκοπήσει πολλές φορές καθυστερημένα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπόρεσαν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να προστατευτούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολλοί οι οποίοι αναφέρθηκαν σε θέματα όπως είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής κτλ. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζω και τα καταγράφω με μεγάλο σεβασμό. Απλώς πρέπει να ξέρουμε το εξή: Σε ένα κοινό έργο όλων των θεσμικών οργάνων που να λαμβάνει υπόψη και τη σημασία της Κομισιόν και των άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίω και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μόνο με τη συνεργασία αυτών των τριών θεσμικών οργάνων μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης, σε μια κοινή συνεργασία για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποια είναι τα διδάγματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τι πρέπει να κάνουμε για μια κοινή και ενωμένη Ευρώπη για την οποία δεν αρκεί απλώς να ονειρευόμαστε, αλλά θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να θέσουμε τα θεμέλια τους και να μπορέσουμε να πούμε στις επόμενες γενιές ότι έχουμε παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην οικοδόμησή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φάιμαν, κύριε Καγκελάριε για τα λόγια σας και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την ιδιαίτερα έντονη και πλούσια συζήτηση. Έχει κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό.